προβώ τρει ανακοινώσει ανακοινώσεις. Πρώτα πρώτα όσον αφορά αποφάσει διαφόρων επιτροπών, ώστε να ξεκινήσουν διοργανικέ ε, διαπραγματεύσει για το, σύμφωνα με το 69 γ όπως αποφασίσαμε ε, την ε, Δευτέρα αρχή της Συνόδου, ζητήθηκαν διάφοροι ε, Έχουν διάφορα αιτήματα τα σύνολο το 69 από το S&D, GUE ε, και από άλλες πολιτικές ομάδες σε σχέση με την Ήτρε που θέλει να ξεκινήσει ε, κάποιες διαπραγματεύσεις επί τη βάση της έκθεσης για τα στατιστικά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και εκεί ήταν η συγκεκριτή του κ.